26 Μαΐου 2016 Liebe Kolleginnen und Kollegen, Αγαπητοί συναδελφοί, με μεγάλη μας ελίπη χτες ακούσαμε ότι ο Τζανλούκα Μπονάνο ε, ξαφνικά απεβίωσε ο συνάδελφος Μπονάνο έγινε ε, στην θητεία του 2014 μέλος της Επιτροπής ε, Βιομηχανίας καθώς και μέλος της αντιπροσωπείας με τις χώρες ΑΚΕ. Ο κύριος Μπονάνο χθες έπεσε θύμα ενός τραγικού τροχαίου και απεβίωσε στη στιγμή. Ήταν επί σειρά ετών ε, δήμαρχος της Πορολίζιας στην Ιταλική κοινότητα, του Ιταλικού Δήμου. Η σύζυγός του επεβίωσε, επιβίωσε και ο κ. Μονάνα αφήνει πίσω του γυναίκα και παιδιά. Αυτή η τραγωδία τάραξε βαθιά πολλούς από εμάς και αυτές τις δύσκολες ε, ώρες θέλουμε να εκφράσουμε την ε, συμπαράστασή μας ε, στην ε, γυναίκα τους, την οποία ευχόμαστε και περαστικά και στην οικογένειά τους. Σας παρακαλώ να τηρήσουμε ενός λεπτού υγιή. vielen dank! Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, τα πρακτικά της συνεδρίασης στις 25 και 26 ε, Μαΐου είναι διαθέσιμα. Δεν ξέρω αν υπάρχουν αντιρρήσεις.